Αποφορά που αφορά την, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν λειτουργεί. Επίτε μας εσείς τι ψηφίζετε, άμα δεν δουλεύει το μηχάνημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η μεταφορά εγκρίνεται με 33 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Et sur la modification Και για την αλλαγή του πίνακα του προσωπικού. Να ψηφιστεί ή όχι. Ωραία λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 35 ψήφοι υπέρ, μία κατά και τρεις αποχές. Την κερδίσατε. Και τώρα... Σχέδιο προϋπολογισμού Πρώτη ψηφοφορία για τη συμφωνία που μας υποβλήθηκε και που συζητήσαμε προηγουμένως. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 24 ψήφοι υπέρ, 9 κατά και 6 εποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική. «24, 9 και 6». Και τώρα τροπολογίες του συγητού. Το σύνολο των τροπολογιών ψηφίζουμε. Alors Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε για τις τροπολογίες του συγκεκριμένου οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη συμφωνία που μόλις εγκρίναμε. On block συνολικά θα τις ψηφίσουμε τις τροπολογίες ή θα τις δούμε μία-μία. Κυρία Γκαρδία Σαμπάλ, έχω χαθεί τελείως. Τι θα ψηφίσουμε τώρα. Τις προφορικές τροπολογίες του συγκητή το πρώτο τμήμα του καταλόγου. Τι. Αυτό που μας μοιράστηκε σήμερα, τι πράγμα. Ή τον κατάλογο. Θα ψηφίζουμε τροπολογία τροπολογία ή τις προφορικές τροπολογίες του εισηγητή που αντικατοπτρίζουν τη συμφωνία. Εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. Έχετε το λόγο να έχω ένα αίτημα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Θα θέλαμε να μην ψηφίσουμε το εδάφιο που διευκρινίζονται όλες οι γραμμές όπου γίνονται περικοπές. Αυτό δεν έχει γίνει ουδέποτε σε έκθεση. Εδώ έχουμε μια γενικόλογη έκθεση και δεν βλέπουμε ποιος είναι ο λόγος να υπάρξει τέτοια ρητή αναφορά σε αυτή την παράγραφο. Αυτό λοιπόν θέλουμε να ψηφεί κατά μόνας. Κυρία Γκαρδιά Σαμπάλ. Λέτε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ειδική μνήμα σε ειδικό εδάφιο των γραμμών που θα έχουν περικοπεί σε σχέση με το σχέδιο προπολογισμού στο σύνολό του. Οπότε Θέλετε να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή ή το πρώτο εδάφιο τέλο πάντων. Ζητείτε η διαγραφή της παραγράφου που λέει ότι στα αγγλικά decrease the level, μείωση του επίπεδου των τακτικών δαπανών. Η πρώτη φράση λοιπόν που λέει decreases the level of the ordinary expenditure υπολογίζεται από το Προεδρείο σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι απαραίτητο, λέει η κυρία Γουάντια Ζάμπαλ, γιατί έτσι και αλλιώ προηγουμένως λέμε ότι υπάρχει ένα όριο στην αύξηση. Οπότε Εγώ προτείνω αυτή την προφορική τροπολογία με βάση την περσινή μου εμπειρία όταν αναφέρονταν όχι μόνο οι γραμμές του περιπλογισμού αλλά και τα αντίστοιχα ποσά. Και αν θυμάμαι καλά χάσαμε αυτή την ε, ψηφοφορία. Γιατί κάναμε αυτό το οποίο τι είναι η κυρία Γκαρθία Σάμπαλ. Τέλο εγώ θα κάνω αυτό το οποίο προτείνει, όπω επιθυμεί. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για το εάν ε, μπορεί να σταθεί στο πλαίσιο της παραγράφου. Εάν η πληρωμή του προϋπολογισμού είναι νομικά δεσμευτική, δεν έχουμε δικαίωμα να αποφασίσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ορίζει το καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. Νομίζω πως το ύψος ε, καθορίζεται με βάση την διαδικασία που αναφέρεται εκεί μέσα και προσαρμόζεται μετά αναλόγως με τα όσα ορίζει το υπηρεσιακό αυτό καθεστώς. Δεν, δεν ξέρω τώρα αν είναι 1,4, 0,8 ή οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι εξαρτάται από το, τον κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση και όχι από το τι θα αποφασίσουμε εμείς. Νομίζω πως δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, εδώ πέρα γράφει 1,4%. Για αμοιβέ κλπ. Euh, euh, ναι κύριε Πρόεδρε, είμαι εισηγητής πέρυσι και είχα ορκιστεί να μην ξαναμιλήσω, αλλά να πω ότι υποστηρίζω το αίτημα της κυρίας Γουάρδια Ζάμπαλ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η αναφορά των συγκεκριμένων σημείων όπου θα υπάρξει μείωση χωρίς να αναφέρουμε στο ποσό της μείωσης δεν έχει κανένα νόημα. Δεν προσθέτει απολύτως τίποτα. Και αν θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτά τα οποία συνέβησαν πέρυσι, έχουν εν τω μεταξύ συμβεί νέα πράγματα. Από τη στιγμή που εγκρίναμε τις προβλέψεις μέχρι τη στιγμή όπου ψηφίσαμε το τελικό ποσό. Γιατί, γιατί εν τω μεταξύ δημιουργήθηκε μια άλλη πολιτική ομάδα. Δεν μπορέσαμε λοιπόν να παραμείνουμε στους ίδιους αριθμούς διότι ήσαν πλέον ανεπίκαιροι. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση της κυρίας Γκουαρδιασάμπαλ είναι η σωστή πρόταση και πρέπει να γίνει δεκτή. Και να πω προς την κυρία Χολμάιερ ότι το ίδιο συνέβη εν πολλής και τον προηγούμενο χρόνο. Είχαμε αποφασίσει πέρυσι ότι για τις τακτικές δαπάνες θα, περιμέναμε, θα περιοριζόμασταν μάλλον στο 1,6. Όταν είδαμε όμως ότι ο πληθωρισμός ήταν αυξημένος και έπρεπε να υπάρξει εκ νέου ρύθμιση, εμείς είπαμε ότι θα μείνουμε στο 1,6 και θα υπάρξουν εσωτερικές αντισταθμίσεις στις διαφορετικές θέσεις. Η πρόταση την οποία προτείνει η κυρία Ζάμπαλ είναι η πιο υπεύθυνη σε δημοσιονομικό επίπεδο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, έτσι ώστε για να μείνουμε στα περιθώρια για την πληρωμή των μισθών το 2006, πληρώσαμε ένα τμήμα των ενοικίων το 16 το 15. έγιναν οι απαιτούμενες μεταφορές στο τέλος του 2015 έτσι ώστε να περάσουμε από ενίκεια του 2015 σε ενίκεια του 2016. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Κοινοβουλίου θα ήθελε το λόγο. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Γενικός Διευθυντής. Μία μικρή διευκρίνηση πάνω στη συγκεκριμένη παράγραφο στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Γουαδιασάμπαλ. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υιοθετηθεί ως έχει η παραγραφός αυτή γιατί λέγεται στα αγγλικά «decrease the level», μείωση του επίπεδου. Ε, όμως εγώ σας κατέθεσα τον προσχέδιο προϋπολογισμού του Προεδρείου που έχει ήδη ενσωματώσει τις περικοπές αυτές. Οπότε έχετε δύο επιλογές. Ή απλά θα λάβετε υπόψη σας ότι η συνδιαλλαγή και το Προεδρείο έχουν προσαρμόσει προς τα κάτω κατά 20 εκατομμύρια ή να διαγράψετε πλήρως την παράγραφο αυτή διότι έτσι και αλλιώς περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και θυμίζω ότι η Κομπή θα υιοθετήσει σήμερα το προσχέδιο επί τη βάση ακριβώς της αρχικής πρότασης. Λοιπόν, ο κύριος ε, εισηγητής μπορούμε να παραμείνουμε μόνο στο πρώτο τμήμα που λέει μείωση της τακτικής δαπάνης για το 17 χωρίς με μία αύξηση εν πάση περιπτώσει κατά 1,4% συγκριτικά με τον προϋπολογισμό του 2016. Να μείνουμε σε αυτή την φράση. Κατάργησε λοιπόν διαγραφή καλύτερα της επόμενης παραγράφου όπως ακριβώς το είναι πρώτη η κυρία Γκουαρδιά Σάμπελ και ε, βοηθήθηκε ως προς αυτό από τον κύριο Ντετρές. Λοιπόν, αφού έγιναν αυτές οι απαραίτητες κωδικοποιήσεις, Έχετε μπροστά σας τώρα τις τροπολογίες του εισηγητή. Για την πρώτη από τις τροπολογίες αυτές, ποιος είναι υπέρ. Α, όχι, πάνε όλα μαζί. Ομαδών λοιπόν για το σύνολο. Διακόπτει πάλι ο Πρόεδρος. Sur l'ensemble de ce texte, qui est favorable Επί του συνόλου του κειμένου αυτού ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι επέχουν. Δεν είναι ξεκάθαρο, θα υπάρξει ε, ονομαστική ψήφος. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Les amendements sont approuvés par 25 voix contre. 26 υπέρ, 13 κατά και 3 αποχές. Δεκτές οι τροπολογίες. Alors, Έχετε τον κατάλογο των ψηφοφόριων μπροστά σας, συνάδελφοι. Έχουμε μία πρώτη προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έχετε τώρα τη συμβιβαστική υπαρίθμου 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 19 υπέρ. Α, για μια στιγμή. Διακόπτει ο πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη, λέγει συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Η συμβιβαστική υπέρ 3 γίνεται δεκτή. Έρχομαι τώρα στην τροπολογία 19. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή, αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. 25 υπέρ 16 κατά. Λοιπόν, συμβιβαστική 4 και 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 23. Υπάρχει κάποιος δισταγμός, διακόπτει την ψηφοφορία ο πρόεδρος. Α, όχι, για το 23 επανέρχομαι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν, έλεγχος δηλαδή ηλεκτρονικός για την 23. Πέρα στις ψηφοφορίες, 23 υπέρ 16 κατά 2 αποχές. Φτάνουμε τώρα στο 29. Όχι, έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική υπαριθμ 6 και είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 7. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ της 7. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 37 υπέρ. Η κυρία Γκουάδια Σάμπαλ έχει ζητήσει πάλι το λόγο. Συγγνώμη που σας διακόπτω για μια ακόμη φορά. Θέλουμε να υπάρξει καταδιέρεση ψήφος εδώ. Γιατί το πρώτο τμήμα της τροπολογίας είναι κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει. Ως εκ τούτου δεν βλέπουμε το λόγο να το υπερψηφίσουμε. Θέλουμε λοιπόν split vote κατά διαίρεση ψήφου. Mais on ne va pas demander au secrétaire général et au bureau de faire une chose qu'on fait déjà. Donc on voudrait faire un split vote. Λοιπόν, από εκεί που λέει ε, ο, ζητάμε από τον Γενικό Γραμματέα να και τα λοιπά. Λοιπόν, ο κ. Ντεπρέ που κατέθεσε την τροπολογία τι πιστεύει. Χωρίς μικρόφωνο ο κ. Ντεπρέ δεν ακούγεται. Νομίζω ότι θα προτιμήσω να διατηρηθεί ως έχει η τροπολογία. Λοιπόν, 37. Ποιοι είναι υπέρ της 37. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή η 37. 38. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 43. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 20 προς 19. Οι 43 και 40 καλύπτονται. Με συγχωρείτε. Δεν ψηφίσατε. Α, ε, να ψηφίζατε. Έγινε η ψηφοφορία τώρα να κάνουμε. Να συνεχίσουμε. 43 και 40. Ενία ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. 43 και 40. 37 votes, 38. Έχω 37 ψήφου. 38 έπρεπε να είναι. Κάποιο λείπει. Τέλο πάντων, πέρασε τη ψηφοφορία. 20 υπέρ, 19 κατά. 44 ε, υπέρ κατέπεσε. 45, 46, 47, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 48. Α, κατέπεσε. 49 καταπίπτει. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, συμβιβαστική 10. Γκαρδία Καρδιαθαμπάλ. Με συγχωρείτε, αλλά. Επειδή δεν είχαμε χρόνο να τα μελετήσουμε, γίνονται τώρα. Χρειάζεται ξεχωριστή ψηφοφορία. Την 53 να την ψηφίσουμε ξεχωριστά της συμβαστικής. λοιπόν, την 53 πρώτα τότε. Πρώτο τμήμα όμως. Πρώτο τμήμα της συμβαστικής 10. 53 κατά προτεραιότητα. Θέλετε να ψηφιστεί το πρώτο τμήμα της 53, σωστά. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα της 53. Herr Uh, Πρέπει να προχωρήσουμε όπως γράφει ο κατάλογος των ψηφοφορίων νομίζω πρώτα τη συμβιβαστική 10 και αν αυτή απορριφθεί να πάμε σε χωριστή ψηφοφορία και να ψηφίσουμε την 53. Σας παρακαλώ λοιπόν ψηφίσουμε πρώτα την συμβαστική 10 και μετά να περάσουμε στην ε, σοφορία κατά τμήματα. Η πρότασή μας είναι το πρώτο τμήμα της 53 της Σοσιαλιστικής Ομάδας να αντικαταστήσει το πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής. Της συμβιβαστικής 10. Dans Στο... βαθμό που υπήρχε συμβασμό, νομίζω λογικό είναι να ξεκινήσουμε από το συμβαστική. Και αν απορριφθεί, να προχωρήσουμε σε αυτό που λέτε. Έχετε το λόγο. Με συγχωρείτε Πρόεδρε, αλλά δεν είναι η στιγμή να αλλάζουμε ό,τι να είναι στι συμβαστικέ. Έχει επέλθει τέτοια ταξία που δεν καταλαβαίνουμε πλέον τι ψηφίζουμε. Μη δημιουργείται νέο αρχιτεκτόνημα τώρα της έκθεσης. Ωραία. Δέκα λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21 προς 17. Δύο εποχές. 11. Συμβαστική 11. Υπέρ. Υπέρ. Για τη συμβαστική 11. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 11. Πέρας. 17-17. Απορρίπτεται, έτσι. 11 λοιπόν, απορρίπτεται. Κύριε Κόρμπελ. Συγχωρείτε, μία σύντομη ερώτηση. Θα έπρεπε να το ξέρω, αλλά ομολογώ ότι δεν ξέρω. Πόσα μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν έχει η Επιτροπή μας, το maximum. <laughs> Mindestens. C'est 41. 41 et euh, on 41. 41. Α, εντάξει. Τώρα το κατάλαβα. Απορρίπτε τη συμβαστική. Κατά συνέπεια, κοιτάζουμε τις, τις τροπολογίες μία-μία. 56, υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται 26 προς 13. Δύο εποχές. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 25 προς 16. Συμβαστική 12, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, συγγνώμη. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Για την 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 21 προς 20. Με συγχωρείτε. 64. Υπέρ. Κατά. 64. You Τι ψηφίσατε υπέρ ή κατά. Μικρόφωνο παρακαλώ, μικρόφωνο. Τι ψηφίσατε. Για την 63 ψήφισα υπέρ. Όχι κατά. Λάθος έκανα. Ε, το αντίθετο, τι να κάνουμε. Εγκρίθηκε, τι να κάνουμε τώρα. Α. Κυρία Χολμάγερ, εψήφισε ε, ψήφισε υπέρ και ήθελε να ψηφίσει κατά. Ε, λάθος έκανε γιατί νόμιζε ότι ήταν άλλη τροπολογία. Ε, κατά λάθος. Το είπε αμέσω. Γι' αυτό ρώτησε αν, μπορεί να ξαναγίνει, αν μπορούσε να ξαναψήσει. Alors, il faut faire un Καλά λοιπόν, τότε θα πρέπει να κάνουμε και ψηφοφορία για να ελέγξουμε για την... Κύριε Πρόεδρε, δεν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός, άρχεται η ψηφοφορία, τελειώνει η πλειοψηφία, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, δεν μπορεί να κολυμπήσει κανείς δύο φορές τον ίδιο ποταμό κτλ. αν κάποιος πιστεύει ότι η ψήφος που έριξε δεν είναι η ψήφος που αρχικά ήθελε να ρίξει, Κύριε Ρούμπιχ, πείτε μας κι εσείς. Κύριε, προτείνω, κύριε Πρόεδρε, προτείνω να ξεκαθαρίσουμε τι έγινε με την 61 και την 62 αν έχει καταπέσει και την 63. Μπορείτε να μου πείτε ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ε, με την 61 τι έγινε. Le 60 a été repoussé. Η 60 απορρίφθηκε. Η 61 εγκρίθηκε. Η 62 δεν ψηφίστη. Θα έπρεπε όμως να είχε ψηφιστεί. Καθότι η 60 απερίφθη, Οπότε 62 δεν κατέπεσε. Διέπραξα μέγιστο σφάλμα. Μην θέτοντας σε ψηφοφορία την 62. Σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Ως εκ τούτου θα ήθελα να ψηφίσουμε την 62 τώρα. Κύριε Φερνάντες, 62, υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικός 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 προς 22. Τρεις αποχές. Έρχεται τώρα η 63. Αυτή έπεται. Ονομαστική ψηφοφορία και εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η 63 απορρίπτεται με 21 ψήφους προς 20. Έπεται 64. Ποιος είναι υπέρ της 64. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71. Κατέπεσε. 72 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 13 προς 20 και 7 αποχές. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20 προς 18 και δύο εποχές. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. 76. Πέρας. Απορρίπτεται. 23 προς 18. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15 εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Διότι δεν σηκώσατε όλο το χέρι. 82. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται με 16 προς 13 και 11 αποχές. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι γίνεται δεκτή δεν είμαι βέβαιος ελέγχουμε ηλεκτρονικά ψηφίζεται την 86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 Τέλος. Απορρίπτεται 21 κατά 20 υπέρ. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Κύριε Γκουαρντια Ζάμπαλ. Θέλατε να ζητήσετε μια καταδιέρεση ψήφων, αλλά Κοιτάξτε, έπρεπε να ζητήσουμε εμείς να τεθεί σε ψηφοφορία η συμβιβαστική. Και ψηφίστηκε η συμβιβαστική. Συγγνώμη. Εμείς ζητάμε να ψηφίσουμε ξεχωριστά ένα τμήμα της συμβιβαστικής. Αυτό γίνεται σε πάρα πολλές εκθέσεις. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες ψηφοφορίας. Όχι βέβαια λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη. Εγώ ζητώ να αφαιρεθεί το τμήμα που ανταποκρίνεται στην τροπολογία 96 του κυρίου Ashworth. εκεί που λέγεται ειδικά με τις δραστηριότητες των Intergroup. Αναφερόμαστε στη συμβιβαστική 16, λέει ο πρόεδρος. Dont on va faire un vote fractionné. Λοιπόν, κατά διέρεση ψήφος. Το πρώτο τμήμα. Σταματάει με τις λέξεις στα αγγλικά interpretation on demand. Λοιπόν, για το πρώτο τμήμα που σταματάμε τις λέξεις on demand, είναι σαφές παρακαλώ. Ε, ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, σας ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Το πρώτο τμήμα γίνεται δεκτό. Το δεύτερο τμήμα σχετικά με τις δραστηριότητες. Ποιοι είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Ποιοι είναι κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής 16 ψηφίζεται. Το δεύτερο τμήμα γίνεται δεκτό 20 ψήφοι υπέρ, 18 κατά και 3 αποχές. Έτσι λοιπόν η συμβιβαστική γίνεται δεκτή. Κάποιος έχει ζητήσει το λόγο. Κανείς. 98. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Λοιπόν, 98 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 100 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 100. δεκτή. 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 102 υπέρ. Α, μάλιστα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 101. Qu'est-ce Merci. Consultation sur le 101. Λοιπόν, 101 ψηφίζεται δεκτή 22 υπέρ 18 κατά 102 ποιοι είναι υπέρ κατά Appel nominal. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 102. L'amendement est repoussé par 24 voix contre 17. Απερίφθη 24 κατά 17 υπέρ. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 108. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται μάλλον, αλλά θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 108. Ψηφίζεται. Απερίφθη. 109. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 110 υπέρ. Κατά. Δεν σηκώνεται όλοι τα χέρια. Ηλεκτρονικός έλεγχος για μια ακόμη φορά. Τέλος. 22 υπέρ 18 κατά μία αποχή. Συμβιβαστική 18. Και εδώ έχει ζητηθεί κατά διέρεση ψήφος για το τελευταίο τμήμα. Το πρώτο τμήμα της 18 και είναι υπέρ. Α, ο κύριος Ντεπρέ θέλει το λόγο. Για το δεύτερο τμήμα, λέει ο κύριος Ντεπρέ, εγώ δεν συμφωνώ με την ιδέα, αλλά στο σημερινό πλαίσιο το να μιλάμε για ανέσεις των βουλευτών είναι πραγματικά ε, τερατοδός υπερβολικό για την κοινή γνώμη να λέμε ότι δεν πρέπει να ταξιδεύουμε κάτω από κακές συνθήκες, αλλά από την άλλη όχι και να λέμε ότι απαιτείται ένα υψηλό επίπεδο άνεση. άνεσης. Λοιπόν, για το πρώτο τμήμα λοιπόν της συμβιβαστικής, εκτός από τη φράση στην οποία αναφέρθηκε και θέλει να καταργήσει ο κ. Ντεπρέ, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, το πρώτο τμήμα γίνεται δεκτό. Το δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής 18. Δεκτό. 21 κατά 17 21 υπέρ, συγγνώμη 17 κατά. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 115. Τέλος. Δεκτή. 27 υπέρ 12. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 117. Τέλος. Απερίφθη 24 κατά 16 υπέρ. 118 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξω. 123 ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 24 προς 16. 124. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. 126 υπέρ. Κατά. Δεν σηκώνετε το χεράκι σα. ηλεκτρονικά. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας. 22 προς 12. 127 υπέρ. Όχι, με συγχωρείτε. Πέφτει. Ε, καταπίπτει. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129 καταπίπτει 230 il est 229 est tombé et alors si 229 est tombé 129 ε, κατέπεσε. Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν έχει εγκριθεί 127. 130. Είναι το ίδιο, είναι η ίδια ψηφοφορία. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Ονομαστική ψηφοφορία για τον 132. Άρχεται η ψηφοφορία. Να Απορρίπτεται το 17 προς 22 δύο εποχές. 133 υπέρ. Κατά. Ε, δεν βλέπω καλά. Δεν είδα τα χέρια σας να σηκώνονται. 133 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται νομίζω. 134 υπέρ. Κατά. Διχασμός. Να επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 20 προς 19 και δύο αποχές. 135 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 136, 137, 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνονται 139, 140, 141 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνονται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 με μία ξεχωριστή ψηφοφορία. Πιστεύετε η χρηματοδότηση για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν πρέπει να αυξηθεί. για αυτήν την προσθήκη του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το υπόλοιπο κείμενο ως ε, 143 ε. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογικέ σκέψει. 1. Υπέρ. Αποχέ. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά να επαληθεύσουμε. Τέσσερα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 20 προς 18 και τρεις εποχές. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 21 προς 17 και δύο εποχές. 6 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απερίπτωται να το επαληθεύσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 προς 25. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 24 προς 12 και 7 αποχές. Φτάνουμε στο τέρμα. Το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται 27 προς 14. Φτάσαμε στο τέλος. Με συγχωρείτε, ήταν κάπως δύσκολα. Αλλά τελειώσαμε. Συνάδελφοι, υπάρχουν άλλα ζητήματα. Δεν βλέπω να υπάρχουν τέτοια. Η επόμενη συνεδρίασή μας, 25 και 26 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Κυρίσω τη λήξη της συνεδρίασης.